Ευχαριστώ κύριε Πέτροπε και έτσι κλείσαμε προσωρινά την συζήτηση για τα ευρωομόλογα. Σας ευχαριστώ και φτάνουμε στην επόμενη συζήτηση αλλά έχω μια αναγγελία από την ομάδα της Σοσιαλιστική ε, να οριστεί ο κύριος Βίστορ Ποστινάν στη θέση του Αρή Μπέρ ε, στην ε, σε σχέσεις ε, της αντιπροσωπείας της Μικτής ε, με την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, συνεπώς ο διορισμός του εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο επόμενο